Συναδελφοί, δεν έχουν προσέλθει πολλοί ακόμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πρέπει να τιμωρηθούν εκείνοι που ήταν στην ώρα τους. Και ως γνωστόν, τιμωρείται αυτός που έχει καθυστερήσει. Επομένως, περνάμε στο σημείο 9 της της διάταξης, παρουσίαση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου 2018 η Κομισιόν ενέκρινε την έκθεση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Τα πορίσματα θα τα μάθουμε σήμερα από τον κύριο Ντελγκάρο από την Γενική Διεύθυνση ΕΡΚ και από τον κύριο Ντόσον από τη Γενική Διεύθυνση Connect η Μπάρμπαρα Γκέσλερ που επρόκειτο να βρίσκεται εδώ δυστυχώς δεν τα κατάφερε γιατί εργάζεται επί του προγράμματος. Εγώ της απάντησα ότι είναι πιο σημαντικό να εργαστεί επί του προγράμματος αυτού για να τελειώσει έγκαιρα παρά να έρθει εδώ και να μας μιλήσει για την ενδιάμεση εξολόγηση. Όμως έχουμε τον κύριο Τελγάδο και τον κύριο Ντόσον που με επάρκεια θα την αντικαταστήσουν στα έγγραφά σας θα βρείτε δύο έγγραφα, την έκθεση, την ίδια, καθώς και το έγγραφο εργασίας. Θα τα μελετήσουμε με προσοχή ως Επιτροπή Πολιτισμού και θα τα λάβουμε υπόψη μας ε, στις συζητήσεις που θα έχουμε για το νέο πρόγραμμα για τη Δημιουργική Ευρώπη. Χαίρομαι πραγματικά για την ε, απόφαση τελευταίας στιγμής της Κομισιόν ε, να παραμείνει αυτόνομο πρόγραμμα το Δημιουργική Ευρώπη. Ήταν ε, σκληρή η μάχη που δώσαμε. Πραγματικά εκνευρίσαμε τους επιτρόπους και τον κύριο Τίμερμανς λέγοντας τους διαρκώς ότι θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να είναι αυτόνομο και στο τέλος ε, πράγματι υποχώρησαν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Μας έκαναν τη χάρη δηλαδή. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στους δύο ε, κυρίους που έχουμε μαζί μας, τους δύο προσκεκλημένους. Παρακαλώ, έχετε μαζί 15 λεπτά. Πώς θα τα μοιραστείτε αυτά, δεν ξέρω. Αλλά έχετε μαζί 15 λεπτά για να έχουμε χρόνο και για τη συζήτηση. Κύριε Ντελγάδο, κύριε Ντόσον, έχετε το λόγο. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρουσιάσω εγώ αυτήν την ε, αξιολόγηση στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Μιλάμε για την διάμεση αξιολόγηση του Creative Europe, της Δημιουργικής Ευρώπης, που ξεκίνησε το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2020. Είμαστε στα μέσα της διαδρομής. Αναφερόμαστε λοιπόν εδώ στην αξιολόγηση αυτή στα τρία πρώτα χρόνια, 2014, 2015 και 2016. Είναι και υποχρέωση από την νομική βάση, άρθρο 18.3, όπου αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο Επιστροπικό Κοινοβούλιο μια έκθεση, μια ενδιάμεση αξιολόγηση ε, από έναν εξωτερικό ανεξάρτητο συνεργάτη. Ε, δεν είναι αυτή η έκθεση βέβαια η παρουσίαση, είναι το πώς η Κομισιόν ερμηνεύει την αξιολόγηση από τον εξωτερικό συνεργάτη. Η επίσημη έκθεση του εξωτερικού συνεργάτη θα δημοσιευθεί σύντομα ε, μιας και έχουμε μια προσέγγιση απόλυτης ε, διαφάνειας. Το Μάιο του 2016 ξεκίνησαν οι εργασίες, ε, χωρίστηκαν σε οκτώ στάδια και ολοκληρώθηκε περίπου τον Σεπτέμβριο του 2017. Είχαμε μια προπαρασκευή, ε, συλλογή δεδομένων, συνεντεύξεις των διαφόρων θεσμικών φορέων, ε, των εθνικών και διεθνών εμπλεκόμενων, μελέτες ε, στον τομέα του πολιτισμού. Υπάρχουν και δύο συγκεκριμένες έρευνες στις οποίες θα αναφερθούμε. Μία για την εποπτεία και μία για το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Είχαμε και ένα παράδειγμα έξι διαφορετικών προγραμμάτων. Έλαβε χώρα μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, μιας και αυτό είναι υποχρεωτικό και βεβαίως στο τέλος είχαμε και τη φάση της ανάλυσης και της ίδιας της σύνταξης της αναφοράς. Λοιπόν, το έγγραφο αυτό μοιράστηκε ταυτόχρονα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση ε, στα μέσα Απριλίου. Έχουμε αυτή την πιο σύντομη λοιπόν έκθεση. Στη συνέχεια έχουμε ένα πολύ πιο πλήρες έγγραφο, το Staff Working Document, όπου μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες των εμπλεκόμενων φορέων ε, πολύ πιο λεπτομερώς, ε, με αριθμητικά στοιχεία και όλες τις πτυχές που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Όλα αυτά αναπτύσσονται εκεί περαιτέρω στο πιο λεπτομερές αυτό έγγραφο. Και τώρα θα αναφερθώ σε δύο κεφάλαια το πρώτο αφορά τα βασικά ευρήματα και στη συνέχεια ε, βεβαίως ε, ποιες είναι οι συστάσεις που προκύπτουν από αυτά τα ευρήματα. Ε, τα ευρήματα πρώτα. Βασιζόμαστε σε έξι κριτήρια τα οποία είναι κλασικά σε όλες τις αξιολογίες της Κομισιόν ε, σημασία, αποτελεσματικότητα, ε, βιωσιμότητα, ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, σε ό,τι αφορά την ε, σημασία, τη σκοπιμότητα δηλαδή. Θέλουμε να προωθήσουμε τη διασυνοριακή ε, κυκλοφορία των έργων, την διασυνοριακή συνεργασία. Θέλουμε οι ε, εταιρείε αυτές οι δημιουργικές να συνεργαστούν μεταξύ τους και αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο και σκόπιμο. Ε, επετέθηκαν οι στόχοι της Creative Europe και ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου της δημιουργίας δηλαδή. Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε ακόμα περισσότερο, να εκμεταλλευτούμε περισσότερο ε, τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται με την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Έχει έναν υπερεθνικό χαρακτήρα ε, ο συγκεκριμένο κλάδος. Τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο επικεντρώνονται εκεί η προσθέμενη αξία του Creative Europe είναι ότι να πτήσουμε ε, υπερεθνικές δράσεις που πολύ σπάνια τη χάνουν υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Η Creative Europe έχει συνεισφέρει σημαντικά έτσι ώστε να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα ε, δίνοντας όθηση στην απασχόληση και εμβαθύνοντας την εσωτερική αγορά μέσω μεγαλύτερης κυκλοφορίας του ε, δημιουργικού περιεχομένου. Θα, θα είχαμε βέβαια πολύ καλύτερα αποτελέσματα με μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Αυτό δεν σας προκαλεί έκπληξη. Η πρόγραμμα, η... Το πρόγραμμα λοιπόν έχει πάει πολύ καλά σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Ο συνάδελφος θα αναφερθεί στα ευρήματα από τα μίντια. Τώρα θα αναφερθώ στο πολιτιστικό σκέλος, στο υποπρόγραμμα το πολιτιστικό το πρόγραμμα έχει, εγγύησεων έχει βοηθήσει στην εφαρμογή του προγράμματος. Είναι ένα νέο στοιχείο του Creative Europe που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Πάνω από 50 εκατομμύρια ε, δάνεια ύψους 5 εκατομμυρίων μπόρεσαν να ε, μοχλευθούν. Ένα σημαντικό έβριμα είναι ότι αυτό που αναφέρουμε ως ε, διατομιακό τομέα εκεί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πραγματικά διατομιακά προγράμματα, δηλαδή προγράμματα, project όπου ε, το medium ε, συνεργάζεται με το πολιτιστικό τομέα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εξέλιξη, όχι επανάσταση αλλά μια εξέλιξη και το γεγονό ότι υπάρχει το Creative Europe αυτό ακριβώ δείχνει ότι θέλουμε να εξελιχθεί το παρόν πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τι συστάσεις, Όπω είπα νωρίτερα, υπάρχει ανάγκη η Creative Europe να αντιμετωπίσει καλύτερα και πιο ισορροπημένα του δύο βασικού στόχου. Ε, πολιτιστική ποικιλομορφία και ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί το σημείο ισορροπία. Ε, θα πρέπει να είναι ποικιλόμορφη αλλά και ποιοτική η ψηφιακή επανάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το δουλέψει περισσότερο. Δεσμευόμαστε λοιπόν να, να αναφέρουμε ετησίως ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο προτείνουμε να συμβεί αυτό στο πρόγραμμα. Στο πολιτιστικό υποπρόγραμμα υπάρχει ανάγκη να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας ε, τους μικρούς ε, εμπλεκόμενους στον πολιτιστικό τομέα. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, σε χρηματοδότηση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και στις ανάγκες τους. Θα πρέπει βεβαίως ε, να γίνει ένα διαχωρισμός μεταξύ των μικρών και των μεγάλων project συνεργασίες. Αυτή τη στιγμή 80% του υποπρογράμματος ε, ε, χωρίζεται σε μικρά και σε μεγάλα προγράμματα, αλλά θα πρέπει να επαναξαλογίσουμε αυτό το διαχωρισμό. Θα επανέλθουμε ε, με συγκεκριμένες προτάσεις επ' αυτού. Θα γίνουν προσπάθειες η ε, Creative Europe και οι διάφορες ε, ατζέντε να έρθουν πιο κοντά η ενιαία ψηφιακή αγορά Παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να έχουν περισσότερε πληροφορίε ε, για τι δυνατότητε συμπληρωματικότητα από άλλε πηγέ χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα είναι έκπληξη για εσά να σα πω ότι μεγαλύτερο μέρο τη υποστήριξη ε, ε, από τα ταμεία στον τομέα του πολιτισμού, τα διαθροτικά ταμεία αλλά και τα ταμεία έρευνα, είναι εκτό Creative Europe και δεν είναι εντό του προγράμματο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι διάφορε πηγέ χρηματοδότηση ό,τι αφορά τα ζητήματα πολιτισμού, για να μπορέσουμε ε, να δώσουμε ε, να έχουμε ένα καλύτερο συσχετισμό, μια καλύτερη διασύνδεση με τις ε, ε, εθνικές και διεθνείς μορφές χρηματοδότησης, θα πρέπει η Creative Europe να βρεθεί στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας. Θα προτείνουμε να ενισχύσουμε το, τα συστήματα ε, πλαίσιο για την ε, παρακολούθηση εδώ στο 2018. Ήδη έχουμε καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και εμπειρογνώμονες σε μια συνάντηση εργασία ε, για να συζητήσουμε την πράξη κατεξιοδότηση όπου θα αποφασιστούν περαιτέρω δείκτε. Οι διαδικασίες υποβολή προτάσεων θα ευθυγραμμιστούν περαιτέρω έτσι ώστε να έχουμε πιο γρήγορη επιλογή. Θα οργανωθούν διασκέψεις για να μπορέσουμε να, διαδώσουμε τα, τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών. Θα πρέπει όχι μόνο να προωθήσουμε τις, ε, τα, έργα, που λαμβάνουν χώρα σε ένα κράτος μέλος, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ένα νέο κριτήριο ε, για τα διάφορα project και τα σχετικά αποτελέσματα. Θα δώσω τώρα το λόγο στο συνάδελφο που θα σας παρουσιάσει το σκέλος που αφορά τα media. Um, σε ευχαριστώ πολύ για το υποπρόγραμμα Media. Θέλω να κάνω την εξή παρατήρηση ότι καταρχάς αφορά και τα κύριο λόγο αφορά τον κινηματογράφο αλλά και τη τηλεόραση και τα βίντεο παιχνίδια και κάθε μορφή, κάθε έργο οπτικό-ακουστικό. Τα κύρια πορίσματα λοιπόν τα εντοπίζουμε στα σημεία προς ενίσχυση, ποιος βελτίωσε. Έχει το υποπρόγραμμα Media λοιπόν συμβάλλει σημαντικά στην ε, ενίσχυση της παρουσίας του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου ως είδου και έχει εξασφαλίσει ένα ρόλο για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο που ξεπερνά την απλή παρουσία του σε μια εθνική ε, αγορά και ως εθνικό κλάδο. Ασχολείται λοιπόν με την ε, διανομή υπερσυνοριακά 400. Βέβαια προσφέρει και στον πολίτη τη μεγάλη αυτή ποικιλία υλικού. Έχει επίσης βοηθήσει τον κλάδο των οπτικοακουστικών να ενισχύσει την κλίμακα δράσης του. Ήταν πολύ περιορισμένη. Θα λέγαμε ένα μπακάλικο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και μικρο επιχειρήσεις. Η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά μπορούν να ενισχύσουν την κλίμακα της δραστηριότητάς τους, σε παραδείγματι με συμπαραγωγές, με κοινή οργάνωση των πόρων τους ώστε να κάνουν μια παραγωγική με μεγαλύτερο προϋπολογισμό και βέβαια διανομή και ορατότητα. Είναι πολύ περιορισμένο ο χρόνος ενώ θα μπορούσαν να τομέα των οπτικοακουστικών και κυρίως την οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες με τις απαιτήσει της για την προαγωγή των ευρωπαϊκών έργων. Για να υπάρχουν ευρωπαϊκά έργα πρέπει και η, ευρωπαϊκή, βιομηχανία ευρωπαϊκός κλάδος, δηλαδή να είναι σε θέση να παράγει τα σχετικά έργα. Τώρα, το ε, προ βελτίωση. Ο Ζωάο είπε ότι είναι πολύ περιορισμένε ε, οι δυνατότητε χρηματοδότηση. Επομένω, ο επιμερισμό. Υπάρχουν και διάφορα ε, διαφορετικά έργα ή σχέδια που είναι οργανωμένα με διαφορετικούς τρόπους αλλά σχετικά άκαμπτους και πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε και να ε, μπορούν να στηριχθούν εκείνα τα έργα τα οποία ίσως να μην ανήκουν αυστηρά στη μία ή την άλλη για να επιτύχουν. Γιατί ό,τι και να λέμε η επιτυχία έχει σημασία στην κινηματογραφική παραγωγή. Συστάσεις. Όπως θα ήταν αναμενόμενο και καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο μισό, καθώς είμαστε στο δεύτερο μισό του προγράμματος, οι συστάσεις είναι ε, διαγραμμικό υλικό, ε, το ίντερνετ έρχεται πρώτο, υπάρχει υλικό που διατηρείται και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Πρέπει να κοιτάξουμε και τη ε, διαγραμμικό υλικό, ε, το ίντερνετ έρχεται πρώτο, υπάρχει υλικό που διατηρείται και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Πρέπει να κοιτάξουμε και τη διαγραμμική κατανομή. Όταν ξεκίνησε το 2013 το Media δεν είχε εμφανιστεί το Netflix στην Ευρώπη. Ενώ τώρα πια έχει καθιερωθεί και διαταράσει ούτως υπήν το τοπίο. Αυτό το λέω σε μια ουδέτερη παρατήρηση, δεν το χαρακτηρίζω ως καλό ούτε κακό γεγονός. Έχει αλλάξει το τοπίο και στο βίντεο on demand, στο VOD, πάλι πρέπει να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις να προλάβουν τις εξελίξεις και να υπάρχει το σχετικό περιεχόμενο. Η ενίσχυση της κλίμακας, η αύξηση της κλίμακας, σύμπεση παραγωγής ουσιαστικά, καθαρά ευρωπαϊκές, ώστε η δική μας παραγωγή να είναι ανταγωνιστική έναντι των μεγάλων αμερικανικών παραγωγών. Ο υποτιτλισμός που θα είναι ένας από τους κύριους τρόπους με, τον οποίο, με τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε την ε, διανομή πέραν των ε, συνόρων και αυτό κοιτάμε να το υποστηρίξουμε και με διάφορα τεχνικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σταματάω εδώ με τα ευρήματά μας. Ευχαριστούμε πολύ και περνάμε στη συζήτηση θα πρότεινα να το ξανακάνουμε με τη διαδικασία ping-pong. Μας αρέσει. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερο στους δύο εκπροσώπους των δύο Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί όντω βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων με πολύ καλά αποτελέσματα. Με χαρά βλέπω ότι έχουμε καλά ε, ε, επιτύχει ως Επιτροπή Πολιτισμού και με την Πρόεδρο κυρία Καμερέφερτ να πείσουμε να διατηρηθεί το πρόγραμμα αυτόνομο. Είναι για μένα πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τον διατομεακό τομέα ε, και ως χώρο πειραματισμού για διατομεακές δραστηριότητες εξελίξεων με βάση συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων, όχι για τα οπτικοακουστικά, όπου βέβαια θέλουμε την ε, ενίσχυση της συνεργασίας με το παρατηρητήριο οπτικοακουστικών, το στοχωρήσουμε. Τρίτη παρατήρηση. Χρήσιμο θα ήταν, πιστεύω, και με ικανοποιεί το γεγονός ότι ο κύριος Δελγάδο μας ε, τουλάχιστον βλέπουμε να έχει περισσότερο δώσει έμφαση στην οικονομική διάσταση και λιγότερο στην ποιότητα την καλλιτεχνική. Ε, μπορώ να κάνω πινκ-πονγκ με τον κύριο Τελγάδο και τις χώρε. και τι συμβαίνει μετά την αποχώρηση της Τουρκίας και πώς συμμετέχουν η Ελβετία και το Ισραήλ. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένε και διαφορετικέ. είναι η οικονομική διάσταση και η διάθεση οικονομικών πόρων για τον πολιτισμό που βλέπω να είναι πολύ χαμηλά. Η μόνη γραμμή δηλαδή που ε, λέτε και μιλώντας ε, για το ειδικό αυτό πρόγραμμα που εμείς έχουμε ζητήσει, ότι υπάρχει ένα Music Moves σχεδιάσει. Ευχαριστούμε. Προσπαθήστε να είστε όσο πιο σύντομος γίνεται. Κύριε Ντελγάδο, κύριε Ντόσον, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Σχεδιάσει. Ευχαριστούμε. Προσπαθήστε να είστε όσο πιο σύντομος γίνεται. Κύριε Ντελγάδο, Κύριε Ντόσον, ποιος θέλει να ξεκινήσει. begin. Θα ξεκινήσω εγώ. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μου δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξω κάποια θέματα. Culture και κάποια διατομιακά προγράμματα. Αλλά πράγματι έχουν διαφορετικά, διαφορετικό αντικείμενο το, το το διατομεακό πρόγραμμα ε, έχει κάποιες ε, ε, εξοχήν διατομεακό χαρακτήρα των προγραμμάτων. Αυτό σχετίζεται όμως με την εξοχήν διατομεακό χαρακτήρα των προγραμμάτων. Αυτό σχετίζεται όμως με την με τη σύλληψη του προγράμματος. Η έναρξη όμως της εφαρμογής του νέου προγράμματος, οι διαπραγματεύσεις που θα προηγηθούν θα, σας, θα μας δώσουν ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε αυτό. Επίσης, να απαντήσω και σε αυτό που είπατε για τη μουσική. Γιατί προφανώς υπάρχει μια προ, φάση η οποία βρίσκεται σε εξήλυση αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα στο πλαίσιο του προγράμματος να, να αναλυθούν δράσεις για τη μουσική. Αξιολογητές ε, συνεκτίμησαν δεδομένα από το 2014, το 2015 και το 2016 από τις συμμετέχουσες χώρες προφανώς και με αυτόν τον τρόπο ε, εξετάσαμε στην αξιολόγηση την νομική βάση που υπάρχει σε κάθε χώρα. Ε, αυτό είναι πολιτική απόφαση και είναι αντικειμενικό. Το, το, το, πρόγραμμα από μόνο του δεν μπορεί να αλλάξει ε, αυτήν την, την προσέγγιση έτσι ξαφνικά χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. ανταγωνιστικότητα και πολιτιστική πυκλομορφία. Πρόκειται για στοιχεία που ενυπάρχουν σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ε, και βλέπω, και αυτό λέει και η εξολόγηση, ότι τα προγράμματα δεν επιλέγονται μόνο με βάση την οικονομική τους αποδοτικότητα. Πάντοτε συνεκτιμάται και η πολιτική ποικιλομορφία κατά την επιλογή και αυτό έχει ε, ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα αυτό να μην ε, χρησιμοποιείται και να μην αξιοποιείται μόνο για την οικονομική αποδοτικότητα. Ε, Βεβαίω αυτά θα πρέπει να τα δούμε και στο τέλος, στην ολοκλήρωση του, του προγράμματος, γιατί λίγα ήταν τα προγράμματα που είχαν ολοκληρωθεί κατά τη φάση της ενδιάμεσης αξιολόγηση. Ε, πάντως ε, η χρηματοδότησή μας ε, μπορεί να αντιμετωπίσει και να αντισταθμίσει ελήψει της αγοράς και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Όσον αφορά τον πολιτισμό, σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι περίπλοκο το θέμα αυτό γιατί ε, υπάρχουν δύο επίπεδα. Όπως είπα, τα ε, συνεργατικά προγράμματα χωρίζονται σε μεγάλα και σε μικρά. Είναι, είπα, τα ε, συνεργατικά προγράμματα χωρίζονται σε μεγάλα και σε μικρά. Είναι κάπως παραπλανητική βέβαια αυτή η διάκριση γιατί υπάρχουν και κάποια μεσαίας κλίμακας προγράμματα. Άλλο θέμα όμως είναι το, το μέγεθος ε, ε των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ε, η πλειοψηφία των φορέων συμμετέχουν σε μεγάλα προγράμματα. Γιατί εκεί κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό γιατί πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία μικροί ε, που χρειάζεται να ε, μεγαλώσουν την κλίμακα των δραστηριοτήτων τους. Μέσα από αυτά τα μεγάλα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με πολύ μεγαλύτερους φορείς και αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για, τις μικρές, για τους μικρούς αυτούς φορείς από το να συμμετέχουν μόνο σε μικρά προγράμματα. Θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό το θέμα και ο συνάδελφος μπορεί να ε, εξηγήσει ε, και τι ακριβώς συμβαίνει με τις ε, ετήσιες διαδικασίες επιλογής. Έχουμε υποβάλει ως Κομισιόν και κάποιες προτάσεις, αλλά θα προβούμε και σε εκτενέστερη ανάλυση αυτής της διάστασης. ναι, τη διατομιακή συνεργασία να σας πω ότι εμείς χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με την DGR. Uh, ναι, για τη διατομιακή συνεργασία. Να σας πω ότι εμείς χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με την DGR ε, για αυτά τα κοινά project ε, στα όρια βέβαια που, του προπολογισμού. Όταν το Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο τροποποίησε ε, τον προπολογισμό και πρόσθεσε ένα εκατομμύριο, Εμεί θα δράξαμε την ευκαιρία και φτιάξαμε από κοινού ένα project για, την πολιτική κληρονομιά, πολυτομιακό, να δείξουμε ε, ταινίε σε αρχιτεκτονικού χώρου, σημαντικού όπω μουσεία ε, που σχετίζονται με την πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης. Ε, ή με έρευνες ή μάλλον ε, σπουδές που να συνδυάζουν την τέχνη και την επιστήμη. Ε, Σύντομα, θα επικεντρωθώ σε ένα θέμα μόνο. Στους ε, συμμετέχοντες στα μικρά, μικρών φορέων που συμμετέχουν σε μεγάλα ε, έργα είναι μεγάλο. Θέλω εγώ να ρωτήσω, οι μικρία έργα αυτά, Είπατε ότι υπήρξαν και κάποια προγράμματα που δεν κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν. Ε, θα με ενδιέφερε να μου πείτε πόσα είναι αυτά τα έργα για τα οποία υπευλήθη η αίτηση, αλλά που δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να χρηματοδοτηθούν. Αριθμό συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω εδώ στοιχεία ε, και λυπούμε. Ίσως όμως να μην εκφράσετε και καλά. Αυτό που είπα δηλαδή νωρίτερα ήταν ότι σε μεγάλο βαθμό οι μικρές ε, όλα τα στοιχεία και θα σας τα αποστείλουμε. Πολύ στο λέει κύριε αυτή η προβολή ακριβώς επειδή είναι μικρά. Παρακαλώ για να απαντήσετε. Κοιτάξτε τα προγράμματα έχουν αυτό το πρόβλημα της ε, θα έλεγα ότι δεν αλλάζει ανάλογα με το ένα μικρή ή μεγάλη επιχείρη, η οντότητα που συμμετέχει. Αλλά θα κοιτάξω και κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά στην αξιολόγηση. Πάντως η, το ποσοστό αποτυχίας υπολογίζω, υποθέτω ότι θα είναι πιο μεγάλο για τις μικρές οντότητες γιατί δεν έχουν τα ίδια μέσα να συμμετάσχουν. Θέτω ότι θα είναι πιο μεγάλο για τις μικρές οντότητες γιατί δεν έχουν τα ίδια μέσα να συμμετάσχουν. με επιτυχία αν δούμε τα βραβεία του παντόρα, της Παντόρας, όπως το Ίντα, οι ταινίες όπως το Ίντα, οι ταινίες του Ken Loach, είναι ταινίες με μικρό προπολογισμό. Ε, αλλά η, ε, ξεπερνάει κατά πολύ την οικονομική αξία, άλλο πολιτιστική αξία, άλλο οικονομική. Έχουμε λοιπόν ένα καλό απολογισμό, ε, μια καλή εμπειρία στην υποστήριξη μικρών ταινιών. Υπολόγισα έτσι 2.000 ε, ε, επιδοτήσεις, αυτό σημαίνει 55.000 ε, σε κάθε επιδότηση. Λίγα λεφτά δηλαδή, στον τομέα του κινηματογράφου, έτσι, γιατί είναι πολύ πιο ακριβή μια ταινία. Ε, βεβαίως μπορεί να είναι αυτή η, η ενίσχυση ταινία. Αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολλοί αναφέρθηκαν στη χρηματοδότηση. Μπορώ να πω... Αυτά τα 60 χρόνια, τα 47, η Πολωνία ε, ήταν υπό την πότα του, του κομμουνισμού. Πολιτιστικά όμως ήταν πάντοτε στην Ευρώπη. Αν είχαμε λοιπόν μια τέτοια ε, εισρωή ε, αμερικανικών ταινιών όλα εκείνα τα χρόνια, ε, όπως έχουμε σήμερα, η, διαταραχή, η διατάραξη ε, της ε, ε, ειρήνης σε εκείνο ένα το ένατο πρόγραμμα. Γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα για τον πολιτισμό. Καθόλου, ούτε ένα. Και δεύτερον, είπατε ότι εξασφαλίζονται μόνο διατομεακές συνεργασίες. Μα γιατί δεν υπάρχει, γιατί είναι τόσο... Θα ρωτήσω και θα του δώσουμε το λόγο. Θα απαντήσω εγώ πρώτος αυτή τη φορά. Συμφωνούμε με αυτό που εκφράσατε, ότι ο πολιτισμός βρίσκεται στην... Το ερώτημα βεβαίως είναι ε, κατά πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε τον, υπο... τον πολιτισμό ε, σε ενωσιακό επίπεδο. Βρισκόμαστε στη φάση προετοιμασία του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Ελπίζουμε τι φιλοδοξίε μας. Για να επανέλθω όμω στο ζήτημα της αξιολόγηση, Πρέπει να σας πω ότι αυτή κατέδειξε ε, ότι δεν υπάρχει κάποιο δίλημα ε, ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και στην πολιτιστική αξία και ποικιλομορφία. Οι δύο αυτές αξίες συμβαδίζουν γιατί ε, όταν μια τηλεοπτική σειρά ή μια ταινία ε, παράγεται μια γερμανική σειρά η οποία παραγεται γερμανικη σειρα η οποια μεταδιδεται ε, σε άλλη χώρα, στη Σουηδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, μεταγλωτισμένη, υποτιτλισμένη. Αυτό είναι πραγματικά μία πρόοδος, ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αποτελεί και, με φέρθηκε ο Ζωάο, συμφωνώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε την διασύνδεση με τα ερευνητικά προγράμματα, με τον ορίζοντα 2020, με τα προγράμματα για το μέλλον της έρευνας. Εγώ δεν θα... και που έχουν και πολιτιστικές εφαρμογές. Και φυσικά υπάρχουν και τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία επίσης παίζουν σημαντικότατο ρόλο και που προσφέρουν τη κατασκευάσει κανείς ε, υποδομές οι οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση του πολιτισμού. Ευχαριστούμε πολύ τον διαπραγματεύσεων για το νέο ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Εμείς άλλωστε ε, έχουμε αναθέσει και την εκπόνηση μιας μελέτης θα το δούμε. Τη μελέτη στις αρχές Ιουνίου, ο κ. Και που, αν κατάλαβα καλά, αποτελεί μια σύνοψη της εκθέσεως. Κάνω λοιπόν ε, μια ερώτηση για να διευκρινίσω. Ξέρουμε ότι έχουν ήδη και μέσα στην εθνική του αγορά τεράστιε δυσκολίε να βρουν χρηματοδότηση, μικρή παραγωγή. Ερωτώ λοιπόν, σε αυτή τη χρονική στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι είναι ο πλούτο μα, πώ μπορούμε να αποφύγουμε απαιτήσει και προσδοκίε τέτοιε όπω αυτό που μα είπατε και μια αντιμετώπιση που αναφέρατε ότι 85% οδηγείται σε αποτυχία και που εν τέλει προοδευτικά και εν τέλει οδηγεί σε αποτυχία όλο το πρόγραμμα. Καταλαβαίνω τη λογική σε διεθνή επίπεδο πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα κανεί να ε, εκφραστεί, να παράγει, να εμφανιστεί και στην εθνική, στην εσωτερική καλύτερα αγορά. Ίσως θα έπρεπε να το δούμε διαφορετικά γιατί ενδέχεται ο κίνδυνος να είναι να κάνουμε όχι ένα βήμα πρόοδου αλλά να αποδυναμώνουμε κιόλα την παραγωγή και δεύτερο πάλι οικονομικού χαρακτήρα γιατί παραμένει το πρόβλημα λέτε ότι εξετάζεται ο συνδυασμό διαφόρων κινδύνευση. Αυτό πώς ακριβώς μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Και μια τελευταία, τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε. Οι δείκτες για τα μέσα μαζική ενημέρωση για τα media, Μπορείτε να μας δώσετε δύο στοιχεία παραπάνω γιατί βλέπω να υπάρχει μια τάση περισσότερο προς τη συγκέντρωση και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να ε, ε, επιδιώξουμε μια συντονισμένη συνεργασία με αυτονομία όμως, με διατήρηση της αυτονομίας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μας έχουν μείνει ακόμα 10 λεπτά και δύο συνάδελφοι. Έχετε εσείς τώρα τη δυνατότητα να δώσετε τις απαντήσεις σας όσο δυνατόν πιο με αυτονομία όμως, με διατήρηση της αυτονομίας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μας έχουν μείνει ακόμα 10 λεπτά και δύο συνάδελφοι. Έχετε εσείς τώρα τη δυνατότητα να δώσετε τις απαντήσεις σας, όσο δυνατόν πιο σύντομα και συγκεκριμένα. Ναι, να προσπαθήσω μετά την κρίση του 2009 ε, να δράσουν σε εθνικό επίπεδο. Όπως είπα στην αρχή, η ιδιαιτερότητα του κρύου με δυσκολία βέβαια από τον εθνικό προπολογισμό. Εμείς έχουμε ως στόχο να στηρίξουμε τις πολιτιστικές είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις παρότι δεν κατάφεραν να λάβουν την επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις παρότι δεν κατάφεραν να λάβουν την επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση την χρηματοδότηση να πει εντάξει δεν χρηματοδοτούμε αλλά τουλάχιστον συνεργάζονται μεταξύ τους αυτοί όχι, δεν λέω αυτό. Απλώς ανακάλυψε ε, ο εξωτερικός συνεργάτης που αξιολόγησε ότι μόνο και μόνο το γεγονός ότι υπέβαλαν και ένα κοινό project ε, κάποιες, αυτό δημιούργησε κάποια λύσουμε το θέμα των εγγύησεων. Εδώ δρούμε σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, Ολο, ε, συμπληρώνουμε την αγορά ως έχει, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις της ε, θέσπισης αυτής της οικονομικής εγγύησης. Εάν η αξία ε, αυτή η οικονομική εγγύηση άλλωστε μας πήρε πολύ χρόνο όσο του θεσπιστεί, δεν είχαμε λοιπόν αρκετά project στη διάθεσή μας για να τα αξιολογήσουμε. Να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο για να συμπληρώσω για την, τα οικονομικά μέσα της εγγύησης ε, στην έκθεση αξιολόγησης όντως αναφέρεται ότι θα εξετάσουμε για το μέλλον ένα μείγμα ε, να υπάρχει ε, και κάποιο όργανο equity για μεγαλύτερα project ε, το λέω αυτό ενδεικτικά διότι εμείς εδώ αυτό το σύστημα εγγυήσεων υποστηρίζει τη δανειοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έγινε μια έρευνα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ ε, δυσκολεύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό. Είναι γνωστό το θέμα αυτό των δανείων. Τώρα από πλευράς equity, επειδή γίνεται μια μελέτη όπου αναλύουμε την κατάσταση, υπάρχει ένα άλλο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο κάποιοι ενδεχομένως μεγαλύτεροι παίχτες, Ευρωπαίοι, με υψηλότερες δυνατότητες ρίσκου και βεβαίως υψηλότερη απόδοση, πολιτιστικοί φορείς, επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αποφεληθούν από ένα σύστημα equity. Να πολλούν μέρος της επιχείρησης, να έρχονται καινούριοι ιδιοκτήτες. Ε, ξέρετε, π.χ. χάρη, το Netflix έχει προπολογισμό δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ το σύστημα εγγυήσεων έχει ένα προπολογισμό 20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Δεν είναι ένα κατάλληλο μέσο λοιπόν εδώ. Τώρα, εάν στα πλαίσια του σχεδίου Juncker αποφασιστεί ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό Netflix, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, λέω αν. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση ξαφνικά που δίνεται. Είναι σαν να φτιάχνουμε ξαφνικά ένα αυτοκινητόδρομο. Εάν βέβαια συμβεί τέτοιο πράγμα. Πάντα όσο πιο σύντομα γίνεται. Σας παρακαλώ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν. Τα είπαν και οι συνάδελφοι, τα είπαν πολύ καλά. Εγώ έχω να πω κάτι πολύ, να ρωτήσω κάτι πολύ απ, λοιπόν στην αξιολόγηση από αυτού. Και κάτι ακόμα, ένα ερώτημα που μπορεί να μην είναι δική σας αρμοδιότητας βέβαια, αλλά πρέπει να το πούμε. Ε, τι θα γίνει στο μέλλον με το Brexit. Εάν δούμε στη Βόρεια Ιρλανδία, στη Νότια Ιρλανδία, στο Κόρκο, στη Σκοτία, στην Ουαλία, ε, τι θα γίνει, ε, ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο όταν έχουμε συνεργασία ε, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στις ταινίε, αλλά και στα, στις εκπομπές, τη απλούστευση και όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τον πολιτισμό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθεί. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Συγγνώμη, Τζούλη, κανονικά ανάποδα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Όπως είπατε, ε, το ποσοστό επιτυχίας ε, είναι πολύ περίπλοκο. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα αυξήσει τον προπολογισμό ή θα σταματήσει τις πρώτες, τις προτάσεις. Ε, αύξηση του προπολογισμού δεν είναι στις δικές μας, δεν είναι δική μας πρόταση. Η μείωση των των, των προτάσεων. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά στο τέλος το ίδιο